επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Έχετε παρατηρήσεις από τα πρακτικά που έχουν ήδη μοιραστεί, τα χθεσινά. Όχι. Οπότε μπορούμε να τα εγκρίνουμε. Έχω και μία ανακοίνωση να σας κάνω.